Αυτές οι διορθώσεις λοιπόν, οι αλλαγές μάλλον, ε, θεωρούνται ε, ε, εγκεκριμένες. Και τώρα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα μιλήσουμε